Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσει στα αρμόδια όργανα, αντιρρήσει δεν βλέπω και διακόπτω τη σύνοδο, την περίοδο συνόδου προς το παρόν.